καλωσορίσω στη συνεδρίασή μα. Θα συζητήσουμε για την περιεγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητώ συγγνώμη που μιλώ αγγλικά, αλλά το υλικό για τον πρόεδρο είναι στα αγγλικά. Έτσι λοιπόν θα μιλήσω αγγλικά. Καλώ ήρθατε στη συνεδρίαση τη επιτροπή ΙΤΡΕ. Λοιπόν, Έχουμε και αναμετάδοση στο διαδίκτυο, έχουμε και πολλούς προσκεκλημένους και σε κάποιους σε αυτό το τομέα είναι ένα θέμα μας απασχολεί εδώ και πολύ καιρό το πρώτο παραπανοπέλο ήταν το 2006 κατά την Αυστριακή Προεδρία. Από τότε έχουμε κάνει πολλά. Το 2007 είχαμε την πρώτη οδηγία για το roaming. Εγώ ήμουν εισηγητής για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαι πολύ περήφανος που μπορεί να προεδρεύσω σήμερα γιατί η αλήθεια είναι ότι ακόμη δεν ε, έχουμε πετύχει απόλυτα την ενιαία αγορά, να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα και τώρα είμαστε ένα χρόνο μετά το τέλος της περιεγωγής. Ξέρετε ότι το Rome Light at Home ήταν ένα σημαντικό βήμα και προς τη σωστή κατεύθυνση. Και έχουμε τώρα και τα άλλα κρατημέλη που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν αυτή τη γραμμή και η Επίτροπος Γκαμπριέλ μας ε, υποσχέθηκε ότι θα κάνει τα επόμενα βήματα. Πρόκειται σαν ε, μαραθώνιο. Μοιάζει με μαραθώνιο. Βέβαια, έχουμε στόχους και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία. Έχει αντίκτυπο στους καταναλωτές. Έτσι λοιπόν, ε, τα επόμενα βήματα για να προωθήσουμε περαιτέρω την ε, ολοκλήρωση στην αγορά τηλεπικοινωνιών είναι σημαντική. Η Επιτροπή Τρία ήταν η Καθήλια αρμόδια επιτροπή και τώρα είμαστε τώρα στην περιεχογή 5 και ελπίζουμε ότι ακολουθείται από το roaming 6 και ελπίζουμε, έχουμε μάλλον μπορέσει να βάλουμε το Roam Light at Home ως ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τις ε, αγορές τηλεπικοινωνιών. Είναι σημαντική η παγκόσμια κινητικότητα και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε θέματα και παγκόσμιας περιαγωγής. Γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι είμαστε κατά μέσο όρο στο 2,5 ευρώ ένα γιγαμπάιτ και το μέγιστο είναι 7 ευρώ. Αλλά αν πάει κανείς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχω πάει στην Κίνα πρόσφατα, είμαστε ε, ακόμη στα 19.500 ευρώ στον επόμενο κόσμο. Και νομίζω πρέπει να δράσουμε. Thanks, uh, who have... Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της ΙΤΡΕ που έχουν εργαστεί για το φάκελο της περιεγωγής, όπως την Πιλάρ, μια Πέτρα, την Αγγέλικα και την κυρία Βαλάν. Ε, Έχουμε προβλέψει ότι η συνεδρίαση μας θα κρατήσει 2,5 ώρε να δούμε αν χρειαζόμαστε όλο αυτό το χρόνο. Οι εμπειρογνώμονε έχουν 15 λεπτά στη διάθεσή τους. Ε, βλέπετε και το ρολόι, εμείς στο Κοινοβούλιο σας δίνουμε πάντα την ευκαιρία να δείτε πώς περνάει ο χρόνος. Λοιπόν, καταρχήν θα ακούσουμε μια εισαγωγική ομιλία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Uh, λοιπόν, νομίζω ότι η πρώτος ομιλητής θα μας μιλήσει για την, ε, τον αντίκτυπο της οδηγίας του Rome Light at Home. Έχουμε τρεις ομιλητές σε αυτό το πάνελ. Θα δώσω καταρχήν στον λόγο στον Τζέρεμι Γκοτφρέι, ο οποίο είναι ο μελλοντικό πρόεδρο τη Μπέρεκ για το 2019 για να μα παρουσιάσει τι γενικέ εμπειρίε με το Rome Light at Home από τη σκοπιά των ρυθμιστών βάσει και των τελευταίων δεδομένων που έχει στη διάθεσή τη η Μπέρεκ, ο φορέα Ρυθμιστικών Αρχών για τι τηλεπικοινωνίε. Το πολύ 20 λεπτά σας δίνουμε. Εμεί υποστηρίζουμε πολύ καλά τον Μπέρεκ γιατί η εναρμόνιση και αμοιβή αναγνώριση θα είναι στα δικά σας χέρια. Σας εμπιστευόμαστε λοιπόν. Εμπιστευόμαστε ότι ο Μπέρεκ αγωνίζεται για την επίτευξη του στόχου να έχουμε μια πραγματική ψηφιακή ενιαία αγορά στις τηλεπικοινωνίες. Το λόγο. Thank you very much, Chair. Um, and I also... Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και για τη στήριξη που μας δείχνετε έχω την αίσθηση ότι πραγματικά υπάρχει καλή συνεργασία έτσι ώστε να επέλθει η εναρμόνιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, οδηγίες και κανονισμοί να ε, οδηγούν προς ε, το ίδιο. Θα, στην ομιλία μου θα υπενθυμίσω το ρόλο της ΜΠΕΡΕΚ στην διασφάλιση εναρμόνισης εφαρμογής του κανονισμού περιεγωγής. Θα αναφερθώ στις ε, υπηρεσίες και στα επόμενα βήματα. Να σας υπενθυμίσω λοιπόν ότι η Μπέρεκ έχει δημιουργήσει δύο σε γραμμές για την περιαγωγή. Έχει σταθεί χρήσιμη στους παρόχους υπηρεσιών, για παράδειγμα, μπορούμε να υπολογίσουμε τα εργαλεία αυτά την ε, δίκαιη χρήση και θεμητή χρήση της περιαγωγής, να δημιουργήσουμε σταθερούς συνδέσμους με τις άλλες χώρες και ούτω καθεξής. Επίσης, ε, καταρτίζουμε εκθέσεις συγκριτικής αξιολόγησης δύο φορές το χρόνο, που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή της ε, περιαγωγής στην Ευρώπη και με θέματα συμβατότητας και στη συνέχεια θα σας ε, παρουσιάσω τα ευρήματα των εκθέσεων αυτών. Επίσης, ε, βοηθούμε την Επιτροπή στην κατάρτιση τιμολογίων, ε, μέγιστον τιμών χρεώσεων κτλ. Συνοψίζοντας λοιπόν, τα αποτελέσματα του Rome Like at Home αναμφίβολα είναι ε, επιτυχημένα. Υπάρχουν στοιχεία που στηρίζουν αυτήν, ε, αυτό το συμπέρασμα. Όλες οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες περιαγωγής και οι περισσότερες ε, χώρες έχουν χρεώσεις οι οποίες μοιάζουν με τις χρεώσεις που κάποιος απολαμβάνει στη χώρα του. Έχουμε δει αύξηση όγκου δεδομένων και κλίσεων από τη στιγμή που εφαρμόστηκε το Roam Like at Home, περιαγωγή σας στο σπίτι σου δηλαδή, είναι βέβαια λίγο δύσκολο να οδηγηθούμε σε έγκυρα συμπεράσματα μετά από μόλις ένα χρόνο λειτουργίας. Όμως υπάρχουν πολλοί πάροχοι λειτουργίας ε, που δεν προσφέρουν υπηρεσίες περιαγωγής και μάλιστα έχουν αφαιρέσει την περιαγωγή από τον ε, τιμοκατάλογο χρεώσεων. Υπάρχουν κάποιε παρεκκλήσει και κάποιε εξαιρέσει. Ευτυχώ είναι μικρό ο αριθμό του και σε γενικέ γραμμέ ε, έχουμε παρατηρήσει μείωση των ε, πωλήσεων χονδρική. Ορισμένε ε, τιμέ μάλιστα είναι πολύ κάτω από το ανώτατο όριο. Μετά, σε ό,τι αφορά την πολιτική δίκαιη χρήση, βλέπουμε ότι περίπου τα τρία τέταρτα όλων των παρόχων υπηρεσιών χρησιμοποιούν μια τέτοια πολιτική είτε σε όλα τα προγράμματα που προσφέρουν, είτε στα περισσότερα, στα τρία τέταρτα. Επίσης, πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούν άλλες διατάξεις του κανονισμού περιαγωγής σας στο σπίτι σου, έτσι ώστε να δημιουργούνται σταθερές συνδέσεις με την ε, χώρα προέλευσης κτλ. Δεν έχουμε βέβαια δεδομένα για τον ακριβή αριθμό των χρηστών που έχουν επηρεαστεί από την εφαρμογή των πολιτικών αυτών. Σε ό,τι αφορά τώρα την κατανάλωση δεδομένων. Σε όλο τον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο η αύξηση είναι πενταπλάσια στη χρήση δεδομένων. Και θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς ε, αν αυτό οφείλεται στον κανονισμό Rome Like at Home ή αν στην ε, γενικότερη αύξηση της χρήσης ε, δεδομένων. Η κατανάλωση δεδομένων ανασυνδρομητή μήνα, αν συγκριθεί με την ανάπτυξη τη... και την αύξηση της κατανάλωσης ε, δεδομένων περιαγωγής, θα δούμε ότι πέρυσι η εγχώρια χρήση αυξήθηκε κατά 20%, η περιαγωγή αυξήθηκε τέσσερις φορές. Η περιαγωγή λοιπόν είναι εκείνη που συνεισέφερε περισσότερο στην αύξηση του όγκου, της χρήσης όγκου δεδομένων. Και η εγχώρια χρήση δεν συνέβαλε τόσο. Αυτό νομίζω πως είναι το πιο αδιάσταστο στοιχείο που έχουμε για τα ωφέλη προς τους καταναλωτές του κανονισμού και πριν την ε, θέση ισχύ του κανονισμού τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Επίσης, μεγάλο ενδιαφέρον έχει, ε, έχουν οι διαφορές στη χρήση των, ε, της περιαγωγής από χώρα σε χώρα. Νομίζω πως αυτές οι διαφορές είναι ενδεικτικές τόσο του τύπου δεδομένων όσο και των χρεώσεων περιαγωγής από διάφορους παρόχους υπηρεσιών. Περνάμε τώρα στα, στον αντίκτυπο του χρόνου κλήσης και του αριθμού των γραπτών μηνυμάτων. Βλέπουμε ότι τα γραπτά μηνύματα διπλασιάστηκαν σχεδόν, καθώς και οι εισερχόμενες κλήσεις αλλά και εξερχόμενες ε, όταν βρίσκεται κάποιος σε περιαγωγή ανέβηκαν ε, στο πενταπλάσιο όγκος δεδομένων επίσης. Και πάλι ε, νομίζω πως είναι εύλογο να συμπεράνουμε ότι όλες αυτές ε, οι αυξήσεις ε, έχουν συμβεί λόγω της θέσης ισχύ του κανονισμού περιεγωγής. Τώρα, το, ο κανονισμός αυτός ήταν πολύ επιτυχημένος στην Ευρώπη. Ωστόσο, η χρέος περιαγωγής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ υψηλέ. εξακολουθούν να είναι υψηλέ. Και εξίσου υψηλέ είναι και οι χρεώσει όταν ξεπεράσει κάποιο ε, τον ε, όγκο δεδομένων ή, ε, ή τα λεπτά που έχει στο πρόγραμμά του. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι πολύ υψηλέ χρεώσει περιαγωγή είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που μόνο έτσι μπορεί να επιληθεί. Περνάμε τώρα στι στις πωλήσει. Βλέπουμε στην ε, μέση ότι υπάρχουν τα γραπτά μηνύματα, αριστερά οι κλήσεις φωνής και δεξιά τα δεδομένα. Η σκούρα μπλε μπάρα αφορά τα χαμηλότερα ποσοστά χονδρικών πωλήσεων που έχουμε παρατηρήσει. Και αφορούν, αφορά αυτά τα στοιχεία που μας έχουν δώσει οι πάροχοι υπηρεσιών. Η γαλάζια μπάρα ε, είναι ο μέσος όρος. Η Ροσβάρα είναι ο υπολογισμός του κόστους ε, που έκανε η Τέρα. Εδώ είχαμε πολύ περιορισμένο αριθμό δεδομένων για να αναλύσουμε και παρατηρούμε ότι πρώτον τα ποσοστά είναι κάτω από τα ανώτατα όρια που βλέπουμε με την κόκκινη γραμμή και μάλιστα αρκετά χαμηλότερα. Ποιο είναι ο λόγος γι' αυτό. Οι τιμέ αυτές ε, είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης ανάμεσα στους ε, παρόχους υπηρεσιών και στους ε, παρόχου χονδρική. Αυτό που παρατηρούμε επίσης, και θα σταθώ σε αυτό στη συνέχεια, είναι πως έχει μειωθεί η διαπραγματευτική ικανότητα ορισμένων παρόχων ε, σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των τιμών. Είναι πιο εύκολο μεταξύ τους οι παρόχοι υπηρεσιών να διαπραγματευτούν και να ε, χαμηλώσουν τις τιμές παρά να διαπραγματευτούν ε, με τον χονδρέμπορο. Επίσης, βλέπουμε τώρα στην διαφάνεια αυτή τον μέσο όρο της τιμής, ε, της χονδρικής τιμής δεδομένων ανά μεγαμπάιτ. Βλέπουμε τα ότι το ανώτατο όριο είναι 0,416 και όχι 0,417. Αυτές είναι οι τιμές που διαπραγματεύτηκαν τα κράτη-μέλη και είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι όλες αυτές οι τιμές είναι πολύ κάτω από το ανώτατο όριο. Ας ε, περάσουμε τώρα στις ε, εξαιρέσεις, στις παρεκκλήσεις. Στις μισές ε, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει καμία τέτοια δυνατότητα, καμία παρέκκληση. Σε ορισμένες άλλες οι εξαιρέσεις έχουν εφαρμοστεί αρκετά. Και μοιράζονται εξίσου σε όλους ε, τους εμπλεκόμενους στις, ε, στη διαδικασία τιμολόγησης. Αυτό εν μέρη διότι έχουν, δεν έχουν καλή διαπραγματευτική ικανότητα στο να ε, καθορίσουν τις τιμές χονδρικής. Σε γενικές γραμμές όμως βλέπουμε ότι αυτές οι παρεκκλήσεις ε, παρατηρούνται σε πολύ μικρούς παρόχους υπηρεσιών. Ορισμένοι MVNOs, ακριβώς επειδή ανταγωνίζονται άλλους ε, παρόχους που προσφέρουν ήδη τις ε, υπηρεσίες Rome Black at Home, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες απόκλησης. Τελικές παρατηρήσεις για τα MNOs και τα MVNOs. Βλέπουμε διαφορές στα έσοδα αναχρήστη. Χαμηλότερη κατανάλωση, ε, αλλά χρήστη τόσο σε εγχώρια χρήση όσο και σε περιαγωγή. Προσπαθούμε να συλλέξουμε όμως δεδομένα ξεχωριστά για την κάθε περίπτωση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα αναλύσουμε. Και ε, τόσο οι νομοθέτες όσο και οι ευρωβουλευτές να έχουν μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, στη συνέχεια η ΠΕΡΕΚ θα συνεχίσει τις εργασίες παρακολούθησης και τον έλεγχο ε, των ε, δεδομένων θα διεξάγει αναλύσεις ε, για το κάθε είδος παρόχου υπηρεσιών ξεχωριστά. Θα προσπαθήσει να αναπτύξει ένα μοντέλο κόστους το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο του κανονισμού στις τιμές και θα συνεισφέρει βοηθώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε στα μέσα του επόμενου έτους ε, να δημοσιεύσει την ε, έκθεσή της. Νομίζω πως ε, δεν χρησιμοποίησα τα 20 λεπτά που είχα στη διάθεσή μου και θα σταματήσω εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ και θα χαρώ πολύ να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση έχετε. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε. Είναι πολύ καλό που βλέπουμε αυτή την διαφάνεια που υπάρχει στις τιμές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι πολύ θετικό γιατί η Μπέρεκ είναι και ένα think tank που είναι μια βασική της λειτουργία. Ξέρουμε ότι η Μπέρεκ όπως και η ΕΙΣΑ για την αγορά ηλεκτρισμού αντίστοιχα ε, είναι επίσης αναγκαία. Αν δούμε την ΕΝΙΣΑ βλέπουμε ότι έχει μεγάλη σημασία να υπάρχει οριζόντια συνεργασία σε αυτό το τομέα, η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί στο μέλλον. Αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το βελτιώσουμε. Είχαμε πολλές διαπραγματεύσεις για την περιαγωγή και η Πέτρα και εγώ ε, στις 4 η ώρα το πρωί είχαμε συζητήσεις για τις ε, τιμές χονδρικής και τώρα οι ανώτερες τιμές που αποφασίσαμε ήταν πολύ υψηλές. Ε, γιατί αν οι τιμές χονδρικής είναι υψηλότερες από τις τιμές λιανικής, αυτό δεν είναι καθόλου κατανοητό. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν η Μπέρκ προς αυτή την κατεύθυνση έτσι ώστε να έχουμε ισχυρή θέση. Θα ήθελα όμως οι βουλευτές να υποβάλουν ερωτήσεις ενδεχομένως και αρχίζουμε ε, με την εισηγήτρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λυπάμαι που έχασα την αρχή, αλλά χαίρομαι που μπόρεσα εστω να παρακολουθήσω το δεύτερο μέρος και παρακολουθώ βεβαίως και τις όλες εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ πέμπτη πρωί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ίδια αριθμητικά στοιχεία όπως χρησιμοποιήσαμε στο νομοθετικό μας εγχείρημα γιατί μιλάμε για τα ε, gigabyte ε, και τώρα βλέπω ότι μιλάμε για ε, gigabytes και εμείς έχουμε στοχοθέτηση την κοινωνία των gigabyte έτσι ώστε οι πολίτες να χρησιμοποιούν μεγάλο όγκο δεδομένων ανάλογα με τις ανάγκες τους. Και αυτό κάνουμε σε κάθε νομοθετικό εγχείρημα. Έχουμε 35 cent ανά megabyte αλλά τι κάνουμε με τα megabyte, ούτε τις ε, χαρτογραφήσεις μπορούμε να διαβάσουμε, ούτε να παρακολουθήσουμε το WhatsApp, ούτε να δούμε ταινίες. Ούτε μπορώ να δω τι συμβαίνει τώρα στην Ήτρε, αν βασιστώ στο 3G με την τιμολόγηση ανά megabyte. Ως προς τους άλλους στόχους, αυτός δεν ήταν ο εύκολος τρόπος για τους καταναλωτές να ταξιδέψουν. Θα πρέπει να δούμε διασυνοριακά τι συμβαίνει και αυτό φορά και τις επενδύσεις για τη χρήση δεδομένων στα κινητά γιατί ο στόχος δεν είναι να παραμένει κανείς στο γραφείο του χρησιμοποιώντας ε, ε, δεδομένα. Θα πρέπει οι καταναλωτές να μπορούν να προωθήσουν και να παρακολουθήσουν και άλλα ή e-health, χάρτες και ούτω καθεξής. Ως προς τις επενδύσεις θα πρέπει να δούμε πώς έχουν προωθηθεί μετά από αυτή την απόφαση, Πολλοί ήταν επικριτικοί για τις ε, χαμηλές ε, τιμές χονδρικής. Ορισμένε χώρες έχουν επενδύσει περισσότερο γιατί υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Πώς είναι δυνατόν σε ορισμένες χώρες να έχετε απεριόριστα δεδομένα και σε άλλες χώρες όχι. Πρέπει να καταβάλλετε ας πούμε 30 ευρώ αντίστοιχα. Άρα θα πρέπει να δούμε τι μπορεί κανείς να αγοράσει με 30 ευρώ. Έχει μεγάλη σημασία να εγκρίνουμε πόσα gigabyte μπορούμε να αγοράσουμε με 30 ευρώ. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες, οι βαλτικές χώρες, Κροατία, Βουλγαρία, ε, Λιθουανία φυσικά, Εσθονία, ε, Λετωνία που έχουν απεριόριστο. Υπάρχει όμως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Πορτογαλία που έχουν πολύ λίγα δεδομένα με αυτή τη τιμή. Και αντίστοιχα άλλες χώρες όπως η Γερμανία που έχουν άλλη αντιστάθμιση. Γι' αυτό θα πρέπει να αναλύσουμε περισσότερο τα δεδομένα και να δούμε πόσο, κατά πόσο μπορούμε να έχουμε πολύ καλές υπηρεσίες κινητής ως προς την αγορά δεδομένων. Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια, γιατί η κυρία Φέρ ήταν αυτή που εκπροσωπούσε τις επιχειρήσεις, γιατί δεν κατέβασε τις τιμές χονδρικής, ενδιαφέρονται να κερδίσουν χρήματα. Αλλά οπωσδήποτε τα έσοδα των Telecom μειώνονται. Αλλά αυτό δεν είναι πλέον επιχείρημα. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Κάρινς. Ευχαριστώ πολύ. Έχω δύο ερωτήσεις. Όλα είναι πολύ ενδιαφέροντα και φυσικά οι καταναλωτές θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα την περιαγωγή. Αυτό επιθυμούν οι πολιτικοί. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω αν έχουν γίνει μελέτες για να δούμε αν υπάρχουν αλλαγές για την, για, ε, για την τιμολόγηση των καταναλωτών χωρίς περιαγωγή. Δηλαδή πώς ε, έχει η τιμολόγηση όταν χρησιμοποιούν τους ε, υπολογιστές στο σπίτι. Ως προς τη, την κερδοφορία των μεγάλων ε, επιχειρήσεων τηλεπικοινωνίας, τι γίνεται σε αυτό το τομέα βλέπουμε ένα μεγάλο κέρδος, αλλά υπάρχουν ίσως και πιο ε, κρυμμένα έσοδα, γιατί βλέπουμε ότι γίνονται μεγάλες επενδύσεις και από τις ε, μεγάλες επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών. Ο κύριος Κόβιτσεκ. Η ερώτησή μου ε, αντικατοπτρίζει αυτά που είπε η κυρία Κουμπάλα Νάτρη, γιατί είμαι Τσέχος πολίτης. Μπορώ να συνεχίσω το γαλλικά αν υπάρχει πρόβλημα με τα τσεχικά. Είναι δική σας η επιλογή. Ε, so, ε, Ευχαριστώ συνάδελφοι. Η κυρία Κουμπάλα Νατρή αναφέρθηκε στο γεγονός ότι σε πολλές χώρες δεν υπάρχει καθόλου πρόσβαση στα δεδομένα και η τσεχική δημοκρατία είναι μία από αυτές τις χώρες. Έχουμε τρεις παρόχους στην τσεχική αγορά, άρα είναι σαφής η αγορά. Έχουν ε, επιμεριστεί την αγορά, την έχουν μοιράσει μεταξύ τους, αν και αρνούνται ότι είναι καρτέλ. Και τα δεδομένα είναι απειροελάχιστα ό,τι καταναλώνετε επιπλέον θα πρέπει να καταβάλετε πολύ υψηλό αντίτιμο. Και επειδή είμαι Τσέχος θα πρέπει να τονίσω ότι 10 χρόνια πριν ο, κύριος Φεραντστοφ, ο προκάτοχός μου, είχε ταχθεί υπέρ της περιαγωγής και μετά τον ε, ε, ε, κυνήγησαν οι αρχές και το πλήρωσε σχεδόν και με τη ζωή του. Εάν χρησιμοποιείτε περιαγωγή με τσεχικό αριθμό, ο τσεχικός πάροχος σας ε, βάζει ένα πολύ ψηλότερο αντίτιμο. Δηλαδή δεν, δεν ισχύει αυτό το Rome Like at Home και οι νομικοί μας σύμβουλοι λένε ότι αυτό είναι απόλυτα δίκαιο. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επίτροπη, γιατί αυτό θα μπορέσει να αρχίσει να συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Δηλαδή, αυτά τα έξοδα ισχύουν όταν βρισκόσαστε στο εξωτερικό ε, περισσότερες μέρες από τις προβληπόμενες. Και δεν μιλώ για την Ελβετία μόνο, όπου οι τιμές περιαγωγής είναι πολύ υψηλές, αλλά γενικότερα και για άλλες χώρες. Οι ψηφοφόροι μου δεν ενδιαφέρονται για οδηγίες. Θέλουν απαντήσεις, σαφείς απαντήσεις. Ε, Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Κοτφρέ και να του ευχηθώ καλή τύχη στα νέα του καθήκοντα. Ξέρω πόσο πολύπλοκο και δύσκολο είναι να προσπαθήσει κανείς ε, ε, να ρυθμίσει όλους αυτούς τους ανεξάρτητους φορείς ε, σε όλη την Ευρώπη. Θέλουμε ένα φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις τηλεπικοινωνίες που να λειτουργεί, καλά. Η περίοδος που έχουμε για να αναλύσουμε τι συνέβη είναι πολύ σύντομη. Παρ' όλα αυτά σας ευχαριστώ για αυτά που μας παρουσιάσετε, γιατί μπορούμε να δούμε μια θετική τάση. Όταν ε, προσπαθείς να ρυθμίσεις κάτι, πάντοτε υπάρχει ένα ερωτηματικό. Θα είναι αυτό κάτι καλό ή όχι και μόνο η ζωή μας δείχνει. Μας δίνει τελικά την απάντηση. Έχω δύο ερωτήσει. Ο κύριος Ρούμπικ ε, ανέφερε τη συνεδρίες που κράτησε μέχρι τις 4 το πρωί και εγώ το θυμάμαι αυτό. Ήμασταν διαιρεμένοι τότε για κάποιες χώρες. Αυτά τα ανώτατα όρια που είχαν τεθεί ήταν πολύ υψηλά, ενώ για άλλες χώρες ήταν πολύ χαμηλά. Έτσι λοιπόν, προσπαθούσαμε να βρούμε τη χρυσή τομή. Και νομίζω ότι περίπου για δύο ώρες προσπαθούσαμε να βρούμε το καλύτερο ανώτατο όριο. Τώρα, να ρωτήσω, βάσει της δικής σας εμπειρίας και βάσει των στατιστικών στοιχείων, υπάρχει βέλτιστο ανώτατο όριο, έχει νόημα να ασκούμε πίεση. Μήπως ε, η πίεση αυτή θα μπορούσε να έχει τελικά αρνητικό αντίκτυπο στην αγορά. Και η δεύτερη ερώτηση. Είχαμε μια αποφασιστική παρέμβαση που έλαβε χώρα και η ερώτησή μου είναι μήπως είμαστε πιο κοντά στο στάδιο οπότε θα πρέπει να αφήσουμε και μόνη της την αγορά, να αφήσουμε ήσυχη την αγορά να λειτουργήσει όπως είπε και ο συνάδελφος, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες ε, οι αγορές. Μήπως ε, θα πρέπει να αφήσουμε τις ίδιες να βρουν ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να λειτουργούν. Πάντοτε ε, τίθεται το ερώτημα, έχει πραγματικά νόημα η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί μπορεί να μην βοηθά πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Ταρέζα Γκρίφιν έχει το λόγο στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που καθυστέρησα, γιατί πολλά συμβαίνουν. Εγώ ως μητέρα, όταν η κόρη μου πήγε διακοπές, για πρώτη φορά ήταν 17 χρονών, ήταν με τους φίλους της και ε, έκανε το υπηκό και της ε, είπα πρέπει τα δικαιώματά σου και γύρισε πίσω με ένα λογαριασμό στο κινητό που ήταν 300 λίρες. Θα έλεγα ότι αυτό δεν ήταν και πολύ δημοφιλές ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πέρα από τις διακοπέ, ε, πολλοί πηγαίνουν στο εξωτερικό και για να δουλέψουν. Όμω θέλω να ρωτήσω τον συνάδελφο για, για το κρυφό κόστο. Το Rome Light at Home ε, είναι πολύ δημοφιλέ στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν μπορώ να λάβω απάντηση αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου <laughs> για το τι θα ισχύσει μετά το Brexit, ε, μετά τα τέλη Μαρτίου. Πώς έχετε απαντήσεις ε, για το ερώτημα αυτό. Γιατί φαίνεται ότι θα συμβεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω μια διαπίστωση και δύο ερωτήσεις. Πρώτον, υπάρχει... Υπάρχει η διαπίστωση ότι θέλουμε ένα ευρώ ανά γιγαμπάιτ. Αυτές τις ε, τιμές θέλουμε να έχουμε και, πρέπει, και αυτό μας δείχνουν οι στατιστικές. Αυτό είναι το καλύτερο για τους καταναλωτές και όλους τους ε, εμπλεκόμενους. Έπειτα, θα ήθελα να μάθω τι άποψη έχετε για τον πληστηριασμό των συχνοτήτων, ε, πώς νομίζετε ότι θα είναι το τοπίο του ανταγωνισμού και ε, τι επιλογές έχει προετοιμάσει η Μπέρεκ ε, σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη. Τι επιλογές έχουν δηλαδή τα κράτη-μέλη για την αγορά γιγαμπάιτ, για την αγορά χονδρικής διότι θέλουμε βέβαια να πιέσουμε την αγορά ώστε να χαμηλώσουν τιμές. Αλλά ποια είναι τα βήματα τα οποία πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις επιθυμίες των πολιτών που έχουμε ακούσει και πολλές φορές από, και από εδώ και όλες, από τους ευρωβουλευτές, για χαμηλότερες τιμές. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα, καταρχάς τα μέλη για τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να τις απαντήσω και το πιο εύκολο είναι τα, το κόστος ευρώ ένα γιγαμπάιτ. Πρώτη ερώτηση. Νομίζω πως είναι ένα πολύ καλό μέτρο για τους τελικούς ε, χρήστες και θα προσέξουμε όταν ξανάρθουμε στο Κοινοβούλιο να σας φέρουμε και τα αντίστοιχα συνοδευτικά στοιχεία. Συμφωνώ μαζί σας λοιπόν. Δεύτερον, ο αντίκτυπος στις επενδύσεις και στις ε, τιμές εγχώριας αγοράς. Νομίζω κάποιος ευρωβουλευτής ανέφερε ότι είναι πολύ δύσκολο μετά από τόσο μικρό χρονικό διάστημα να κάνουμε μία απλή αξιολόγηση της κατάστασης. Συμφωνώ. Μία δυσκολία υπάρχει στην αξιολόγηση του αντικτύπου στις επενδύσεις στις ε, χώρες τιμές. Να, μπο, να ξέρουμε δηλαδή να, τι θα είχε γίνει εάν απουσίαζαν αυτές οι χρεώσεις περιεγωγής, αυτές ο κανονισμούς. Δεν έχουμε αναλύσει επίσης την περίπτωση των συγχωνεύσεων όταν, για παράδειγμα, σε μία αγορά συγχωνεύονται δύο πάροχοι υπηρεσιών και ενώνουν τις δυνάμεις τους. Χρειαζόμαστε εμπειρία από αγορές που έχει συμβεί αυτό. Να σας υπενθυμίσω όμως ότι χρειάζεται τεράστια προσπάθεια και τεράστιος όγκος δεδομένων που έπρεπε να συλλέξουμε έτσι ώστε να γίνει αυτή η ανάλυση. Τώρα θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε τις ε, διακυμάνσεις ε, στις ε, εγχώριες τιμές μετά από λίγο καιρό, όταν θα έχει οριμάσει κάπως η αγορά. Οι επενδύσεις είναι πολύ δύσκολο να αναλυθούν και να μπορέσουμε να κάνουμε μια συσχέτιση ανάμεσα στον κανονισμό και στις επενδύσεις σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Νομίζω πως δεν έχουμε μέχρι τώρα στοιχεία συσχέτισης ποιότητα των υπηρεσιών και των ε, τιμών, ακριβώς επειδή είχαμε τεράστιο όγκο δεδομένων να αναλύσουμε. Μετά, έγιναν κάποιες ερωτήσεις για την εγχώρια τιμολόγηση και γιατί ορισμένες αγορές έχουν, για παράδειγμα, με 30 ευρώ απεριόριστο όγκο δεδομένων και άλλες ε, χώρες τελείως διαφορετικό σύστημα τιμολόγησης. Νομίζω η Ιρλανδία είναι μία από αυτές τις αγορές όπου ένας πάροχος ε, προσφέρει απεριόριστο όγκο δεδομένων. Νομίζω πως αυτό έχει να κάνει με τις δυνάμεις του ανταγωνισμού στην κάθε αγορά. Ε, και δεν θεωρώ ότι το «Rome Like at Home έχει επηρεάσει καθόλου το τοπίο εκεί. Ε, η αγορά καθορίζεται από τον αριθμό των παρόχων, από τον αριθμό των MVNO, ε, από, άλλες, ε, από άλλους παράγοντες. Τώρα, οι διαφορές από αγορά στην αγορά είναι είναι ένα γεγονός, ακούσαμε για το τι συμβαίνει στην ε, Τσεχοσλοβακία, όμως αυτό θεωρώ πως ε, πρέπει να εξεταστεί από τους ε, ίδιους τους Τσέχους, έτσι ώστε να διαπιστώσουν αν έχει γίνει κάποια παρέμβαση και να την χειριστούν. Μετά, στην περίπτωση προτινόμενων συγχωνεύσεων είναι πολύ σημαντικό η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ε, Κομισιόν να ε, διεξάγει μια ανάλυση για το αν, ε, ο, για το αν έχει γίνει προκήρυξη κτλ. για το αν αυτές οι συγχωνεύσεις επιτρέπεται να γίνουν. Μετά, υπάρχει, τώρα, υπάρχουν όρια στις τιμές εχονδρικής, αν αυτές θα αλλάξουν, αν μπορούν να πιεστούν προς τα κάτω, όπως ε, ακούσαμε, η εμπεριστατωμένη απάντηση προαπαιτεί μία σε βάθος κατανόηση του κόστους που βρίσκεται από πίσω από αυτό που βλέπουμε. Η ανάλυση μας βασίζεται σε δεδομένα μια συγκεκριμένη χρονική βασιζεται σε δεδομενα μια συγκεκριμενη χρονικής ε, περιοδου και μια συγκεκριμένη ε, στιγμή. Έχουν αλλάξει από τότε Νομίζω πως αυτό που χρειάζεται είναι να γίνουν πιο... να, έχουμε περισσότερη εμπιστοσύνη στα δεδομένα που συλλέγουμε και στην ικανότητα ανάλυσης. Το θέμα είναι ότι πρέπει να, καλύψουμε, πρέπει να καλυφθεί το κόστος της πρόσθετης ε, κίνησης δεδομένων. Και εδώ ίσως δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα κρατημέλη και στα δίκτυα υπηρεσιών. Βέβαια, οι διαφορές έχουν να κάνουν με τον πληθυσμό μιας χώρας, με την ε, κατανομή του πληθυσμού, ε, με την ε, γεωγραφία μια χώρας και, με διαφορούς, και από διάφορου άλλους λόγους. Νομίζω πως όσο περισσότερες και καλύτερες πληροφορίες που έχουμε για το κόστος, τόσο καλύτερα θα μπορέσουμε να δούμε το θέμα των ανώτατων ορίων. Νομίζω πως δεν είναι δουλειά μας να παρεμβαίνουμε στην αγορά και να ρυθμίζουμε να τη ρυθμίζουμε. Υπάρχει ένα πλαίσιο πίσω από αυτόν τον κανονισμό και άλλους σχετικούς κανονισμούς, το οποίο θεωρεί ότι η παρέμβαση πρέπει να γίνεται μόνο όταν ε, η αγορά έχει, κάποια, έχει κάποιο πρόβλημα. Οι χρεώσεις για την ε, περιαγωγή δεν μας δείχνουν ακόμα πώς ε, έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πώς ε, έχει πρόβλημα η αγορά. Έχει αποτύχει. Ούτε και πώς οι χρήστες δεν έχουν καταφέρει να υπολογίσουν το πραγματικό κόστος ε, της περιαγωγής. Ίσως ο κανονισμός Roam Like at Home να μην είναι η πιο κατάλληλη παρέμβαση, όμως τα αποτελέσματα που ε, επιφέρει για τους τελικούς χρήστες είναι πολύ καλύτερα από ό,τι προηγουμένως. Μετά με ρωτήσατε τι θα γίνει μετά το Brexit, με την παριαγωγή. Αυτή την ίδια απάντηση έχω και εγώ. Αυτό θα εξαρτηθεί από το τι Brexit θα έχουμε. Και δυστυχώς ε, δεν έχω μαντικές ικανότητες ε, αρκετές έτσι ώστε να απαντήσω αυτή την ερώτηση. Ναι, σχόλιο εκτό μου του κοροφώνου από τον κύριο Ρίμπιγκ. Κύριε Πρόεδρε, εσεί νομίζω κάνατε μια ερώτηση για τις συχνότητε και τι θα γίνει εκεί. Δεν είμαι ακριβώ σίγουρο που θέλατε να καταλήξετε. Σε ό,τι αφορά την κατανομή του φάσματος συχνοτήτων, ε, κάποια κρατημέλη έχουν ε, αναθέσει συγκεκριμένο φάσμα για τα 700 MB ε, και για άλλες συχνότητες. Αυτή η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί τα επόμενα χρόνια. Ορισμένα χρόνια, ορισμένες χώρες θα ανοίξουν την αγορά τους, ορισμένες ε, θα δουν αυξήσεις στις χρεώσεις. Βλέπουμε ότι αυξάνεται πολύ η χρήση όγκου δεδομένων. Και για να ανταποκριθούμε στις ε, απαιτήσεις της αγοράς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία 5G η οποία μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να διακινεί μεγάλο όγκο δεδομένων με χαμηλότερο κόστος, ε, αλλά χρειάζονται, χρειάζεται να τις ε, αναταθούν οι αντίστοιχες συχνότητες. Αυτό βέβαια είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών η ανάθεση ραδιοφάσματος. Και νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας, έχουμε πολλά να μάθουμε. Ήδη σε αναπίσημο επίπεδο γίνονται κάποιες ανταλλαγές πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών. Νομίζω πως μας έχει υποφελήσει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλή απαρχή της συζήτησης. Τώρα φτάνουμε στη δεύτερη ε, σειρά. Ε, ως προς αυτά που είπε ο Κάρινς, ε, η Μπέρεκ δεν είδε τι γίνεται με τις εγχώριες τιμές ως προς την επεξεργασία ε, ανώτατων τιμών για την περιαγωγή. Όχι, ακόμα δεν έχει διενεργηθεί αυτή η μελέτη. Νομίζω ότι θα μας απασχολήσει στο μελλοντικό πρόγραμμα της Μπέρεκ. Θα πρέπει όμως να έχουμε περισσότερη πείρα, γιατί είναι πολύ δύσκολο για μας να προβλέψουμε ποια θα είναι η πορεία των εγχώριων παρόχων ε, λήψη περιαγωγής. Υπάρχουν παροχοί οι οποίοι ε, προσφέρουν πακέτα που δεν ε, περιλαμβάνουν την περιαγωγή και υπάρχουν ε, πάροχοι που έχουν αποσύρει την περιαγωγή από τα πακέτα. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει εμπεριστατωμένη μελέτη για την παροχή υπηρεσιών στην περιαγωγή. Δεν έχουμε όμως τα στατιστικά δεδομένα. Τώρα περνάμε στο δεύτερο μέρον τι γίνεται με την ε, επίπτωση του Rome Like at Home. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Λίζα Φιούρ που είναι Γενική Διευθύντρια του, ε, της ΕΤΝΟ που είναι η Ένωση Ευρωπαϊκών Φορέων Εκμετάλλευσης Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων αλλά και της ΕΣΚΟ. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε ακούσουμε από εσάς ποιες είναι οι επιπτώσεις στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ρούμπιχ αλλά και τον ε, πρόεδρο της ΙΤΡΕ, τον κύριο Μπούζεκ, που μας ε, καλέσατε για να μιλήσουμε σε αυτό το φόρουμ. Δεν θα μιλήσω για την έξω που αφορά το θέμα της ασφάλειας, αλλά την έθνο και τα μέλη της. Επίσης, Ευχαριστώ τον κύριο ε, Godfrey και τους ευρωβουλευτές γιατί μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό και ορατό θέμα έμπρακτα. Εγώ είμαι Γενική Διευθύντρια της ΕΤΝΟ που είναι ο βασικός ευρωπαϊκός φορέας εκμετάλλευσης των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Όλα τα μέλη μας είναι επιχειρήσεις που κάθε χρόνο επενδύουν στα ψηφιακά δίκτυα της Ευρώπης, η T-Mobile, η Telefonica, Orange, Proximus και TIM, για να αναφέρω μόνο μερικά από τα μέλη μας. Και πριν μιλήσω επί της ουσίας του θέματος που μας απασχολεί σήμερα, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι επιχειρήσεις μας ασχολούνται ιδιαίτερα με συγκεκριμένα θέματα. Όπως ε, είπαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η βασική μας προτεραιότητα είναι να εξασφαλίσουμε τους, ε, στους πολίτες και τις επιχειρήσεις τεχνολογίες εχμής. Άρα όλες οι επιχειρήσεις μας θέλουν να δημιουργήσουν νέα δίκτυα οπτικών ινών και φυσικά να εκινήσουμε το δίκτυο 5G. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη μας είναι ε, επικεφαλής του 70% των επενδύσεων σε τεχνολογίες εχμής και ο τομέας συλλογικά επενδύει 49 δις ευρώ για νέα δίκτυα, υπηρεσίες και εξοπλισμό. Αναφερθήκατε στο γεγονός ότι ο ανταγωνισμός είναι παγκόσμιο σήμερα και καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ζωτικής ε, σημασίας, όχι μόνο για το μέλλον των τηλεπικοινωνιών, αλλά αυτό που μας ε, ενδιαφέρει είναι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και ο ευρωπαϊκός ανταγωνισμός. Αν δούμε το Rome Like at Home, θέλουμε να λάβουμε υπόψη την πείρα των παρόχων στην εφαρμογή του Rome Like at Home γιατί στο τέλος οι λιανικές τιμές ήταν μια συνολικά επιτυχής διαδικασία. Οι καταναλωτές και οι πελάτες ε, ανταποκρίθηκαν πολύ καλά στο Rome Like at Home. Και μια ένδειξη είναι ότι όσον αφορά τα μέλη της έτνο, υπήρχε μία πολύ καλή μετάβαση και ασφαλής μετάβαση τη χρήση δεδομένων στην Ευρώπη. Ο κύριος ε, ε, Godfrey μίλησε για αυτό το θέμα από την Μπέρεκ. Θα πρέπει όμως να δούμε τι συμβαίνει αυτό για όλες τις επιχειρήσεις. Έπρεπε να κάνουμε μια μεγάλη επένδυση σε ένα ιδιαίτερα μικρό χρονικό διάστημα. Υπενθυμίζω στους ανθρώπους ότι τη στιγμή που δεν καταβάλουμε κόστος περιαγωγής γίνεται μια μεγάλη εργασία σε επίπεδο παρόχων. Δηλαδή αυτός ο όγκος εργασίας παραμένει χωρίς αντίτιμο και κανένας πάροχος ε, δεν διαθέτει δίκτυο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή δεν υπάρχει αντίτιμο για την περιαγωγή, αλλά θα πρέπει να έχουμε ολόκληρη την υποδομή έτσι ώστε οι καταναλωτές να έχουν τις δωρεάν αυτές υπηρεσίες. Και αυτό σημαίνει μία τάχιστη προσαρμογή του συστήματος όλων των παρόχων και ήταν ένα ογκώδες εγχείρημα από εμπορικής και τεχνικής πλευράς. Και είμαι πολύ υπερήφανη διότι ε, πήγε πάρα πολύ καλά για όλα τα μέλη της ΕΤΝΟ. Χαίρομαι επίσης ιδιαίτερα γιατί από θεσμικής πλευράς αναγνωρίζεται αυτή η εργασία γιατί οι επιχειρήσεις Telecom συνεισέφεραν άμεσα στην επιτυχία των μέτρων τύπου Rome Like at Home. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα ερωτήματα για το παρόν, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο ε, υπάρχει ένας κελισμός, ε, κατά πόσο δηλαδή θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω επενδύσεις από όλη την επενδυτική κοινωνία, αλλά θεωρώ ότι η πάροχοι πάντα θα είναι μέρος της λύσης, όχι μέρος του προβλήματος. Αν δούμε το ε, μεγαλύτερο πεδίο των ε, τηλεπικοινωνιών βλέπουμε ότι υπάρχουν ελάχιστες εξαιρέσεις που ζητήθηκαν ή χορηγήθηκαν, κάτι το οποίο δείχνει ότι οι κανόνες λειτουργούν και λειτουργούν πολύ καλά. Αναφέρθηκα σε αυτό ειδικά γιατί για μας και για τις επιχειρήσεις η σταθερότητα και το βάσιμο το να μπορούμε να βασιστούμε στα δίκτυα ε, έχει μεγάλη σημασία μέσα στα πλαίσια του 5G το οποίο επίκειται. Κανένας επενδυτής δεν χαίρεται όταν ε, του πούμε ότι δεν θα έχει έσοδα από την περιαγωγή. Πέρα από τους ε, λιγότερους πόρους, για, την, ε, για τις επενδύσεις έχει μεγάλη σημασία η νομική ασφάλεια. Και γι' αυτό το λόγο θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις ρυθμιστικές αρχές για την εφαρμογή των κανόνων αποδοτικά και με σταθερό ευεργέτημα του καταναλωτή. Ξέρω ότι τα μέλη έχουν ε, διαβλέψει ορισμένες απάτες και τους κανόνες σε σχέση με την ε, δικαιοχρησία. Γι' αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε τον κανονιστικό διάλογο και να έχουμε μία πραγματιστική εφαρμογή των κανόνων. Έχω τέσσερα μηνύματα ε, υπομορφή συγκεφαλαίωσης, δεν έφερα διαφάνειες, απλώς ε, κάλυψα αυτά που ήθελα με την ομιλία μου. Η Ευρώπη θα πρέπει να έχει τα καλύτερα δίκτυα στις καλύτερες τιμές, έτσι ώστε ολόκληρη η ε, Ήπειρος να μπορεί να συμβαδίσει με, την, με τους παγκόσμιους ανταγωνιστές. Δεύτερον, το Rome Like at Home κατέβαλε μεγάλη ε, προσπάθεια και τα ευρωπαϊκά δίκτυα ήταν αναπόσπαστο μέρος αυτής της λύσης και της γενικότερης αποδοτικότητας. Τρίτον, σταθερότητα και ασφάλεια ως προς τους κανόνες μας. Αυτό είναι ύψης της σημασίας, ιδιαίτερα για μια ευαίσθητη στιγμή ως προς το επενδυτικό κλίμα της Ευρώπης. Τέταρτον, όλα τα μέλη και η έτνο... Είμαστε στη ε, διάθεση των ε, εθνικών παρόχων της ΜΠΕΡΕΚ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να συνεργαστούμε επί των ε, εξελίξεων σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στον επόμενο ομιλητή, ο κύριος Μιχαήλ Κράμερ, ο οποίος είναι διευθύνων εταίρος στη Βεντοκομ και θα μπορούσε να μας παρουσιάσει τις ε, κοπιά ε, των ε, MVNOs, δηλαδή των φορέων τηλεπικοινωνίας για τα ιδεατά δίκτυα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Μικρόφωνο παρακαλούμε. You can, ah, it works now. Okay. Uh, thank you for the... Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι εξαιρετική ευκαιρία Είμαι εδώ για να σας ε, παρουσιάσω την άποψη ενός ε, ε, μικρού φορέα τηλεπικοινωνιών ιδέα του δικτύου που δραστηριοποιείται στην Αυστρία σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές αγορές. Η προσωπική μου εμπειρία είναι 20 ετών ε, σε αυτό τον κλάδο ως διευθυνός σύμβουλος ε, σε εταιρείε εμενός όπως ε, η Orange και η TNI e Plus στη Γερμανία. Ξέρω πολύ καλά λοιπόν τον κλάδο και την ανάπτυξη του Ρόμιν και συζητάμε χρόνια το θέμα αυτό. Καταρχήν, θέλω να κάνω μια σύντομη εισαγωγή για την εταιρεία που έχω ιδρύσει. Ιδρύσαμε μια εταιρεία μέσω μετά την ε, συγχώνευση της Orange και της Hatch στην ε, Αυστρία. Εδώ έχουμε το αποτέλεσμα ενός καθεστώτος διορθωτικού για τη συγχώνευση. Ιδρύσαμε την εταιρεία το 2013 και αρχίσαμε να λειτουργούμε στην Αυστρία τον Ιανουάριο του 2015 και στη Σλοβενία τον Μάιο του 2017 και φτάσαμε ένα μερίδιο της αγοράς στην Αυστρία 6,5% μέσα στα 3,5 χρόνια και στη Σλοβενία μέσα σε ένα έτος 2%. Είναι αξιοσημείωτο αυτό γιατί πρέπει να έχετε κατά νου ότι πάνω κάτω είμαστε ειδική εταιρεία, δηλαδή λειτουργούμε μόνο στην αγορά των καταναλωτών δεν προσφέρουμε λύσεις ε, για, τους, για τις επιχειρήσεις και για την Αυστρία. Ε, είμαστε, έχουμε μια πολύ σημαντική αγορά, η μεγαλύτερη αγορά για τους ε, καταναλωτές ηλιανικές που χρησιμοποιούν τα smartphone τους. Έχει ανέβει ήδη το μερίδιο της αγοράς μας σε αυτούς κατά 10%. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό σε μια ανταγωνιστική αγορά. Πρόκειται για μια μοναδική πρόταση που προσφέρουμε ε, ως εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, ε, γιατί υπασχόμαστε πλήρη διαφάνεια και δικαιοσύνη και η πρότασή μας είναι να μην αυξήσουμε ποτέ τις τιμές και αν βελτιωθούμε ή γίνουμε φτηνότεροι, αυτό αυτόματα γίνεται για όλους τους πελάτες μας. Οι πελάτες λοιπόν ε, δεν χρειάζεται να ασχολούνται ε, με το να αλλάξουν ε, τιμή, αυτόματα μεταφέρονται στην καλύτερη προσφορά και γι' αυτό μπορέσαμε να έχουμε αυτομερίδιο της αγοράς σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Έχουμε αντίκτυπο στην αγορά. Στο γράφημα αυτό βλέπετε το δίκτυο τιμολόγησης από την Εθνική Ρυθμιστική Αυστριακή Αρχή. Και βλέπετε εδώ διάφορα βήματα. Καταρχήν, αυξήθηκαν οι τιμές στην Αυστρία μετά την συγχώνευση των δύο εταιριών, της Χάτσας και της Όραντς. Βλέπετε εδώ ότι η μέση τιμή αυξήθηκε από 83 σε 104. Και όταν ε, ξεκινήσαμε ε, με την ε, κύρια εταιρεία μας στην αγορά με τη HOT το 2015, ξανά πέσαν οι τιμές γιατί πριν είχαμε χαμηλό ανταγωνισμό. Όταν εισηγάγαμε όμως εμείς τη HOT μειώθηκαν οι τιμές Ήμασταν δηλαδή μια ισχυρή δύναμη στον ανταγωνισμό και εδώ αποδεικνύεται αυτό όχι μόνο από την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή αλλά και από την Εθνική Αρχή Ανταγωνισμού της Αυστρίας. Ε, το αναφέρω αυτό όχι μόνο γιατί είμαι περήφανο για αυτό το αποτέλεσμα αλλά επειδή ε, υπάρχει ένας κίνδυνος απέναντι στη θέση αυτή λόγω ε, του καθεστώτος περιαγωγής ε, για τις τιμές χονδρικής. Ίσως να μην γνωρίζετε, αλλά κυκλοφορούν κάποιες φήμες ότι αυτή η αύξηση της χρήσης του Ρόμπιν δεν είναι και τόσο τεράστια. Σας δείχνω λοιπόν αυτά τα μοντέλα της χρήσης. Κυκλοφορούν θύμες ότι ότι είναι ουσιαστικά ένα αποτέλεσμα τους καλοκαιρινού μήνες. Για να δούμε όμως τώρα εδώ ποιο είναι το αποτέλεσμα. Το πρώτο, ο πρώτος αντίκτυπος στους καταναλωτές είναι ότι υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που χρησιμοποιούν την περιοχή στο εξωτερικό και το μοντέλο της χρήσης επίσης αλλάζει και αυξάνεται. Για να δούμε τους χρήστες. Εδώ Βλέπετε την εικόνα της HOT που έχει πάνω από 80.000 συνδρομητές. Βλέπετε ότι ο αριθμό των χρηστών που χρησιμοποιούν υπηρεσίε περιαγωγή εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί ε, επί δύο. Και επίσης για να απομακρύνουμε και την φήμη e e, ότι οι πελάτε MVNO δεν χρησιμοποιούν τόσο πολύ τι υπηρεσίε roaming. Το 70% των χρηστών χρησιμοποιούν την περιοχή τουλάχιστον μία φορά ετησίω. Και βλέπετε εδώ ότι δεν έχουμε εποχικότητα στην αύξηση των χρηστών. Αυξάνεται ακόμη περισσότερο τους μήνες που δεν έχουμε διακοπές. Τι γίνεται με τα λεπτά, λοιπόν, ένα χρήστη. Λοιπόν, τα λεπτά ομιλίας, γιατί όλοι μιλάνε για τα δεδομένα. Αυξήθηκαν τα λεπτά ομιλίας κατά μέσο όρο επί πέντε πριν από το, σε σχέση με το πριν το Rome Lab at Home ε, και έχουμε υψηλότερη αύξηση τους μήνες όπου δεν έχουμε διακοπές. Πάλι εδώ δεν έχουμε εποχικό αντίκτυπο. Και πάλι εδώ βλέπετε ένα εντυπωσιακό γράφημα για τα δεδομένα. Η κατανάλωση των δεδομένων ε, πραγματικά εξεράγει, δηλαδή σχεδόν επί 45 μετά το Rome Late at Home και έχουμε και αύξηση τους κανονικούς μήνες παρά τους ε, τυπικούς ε, μήνες που χρησιμοποιείται η περιεγωγή, της διακοπές δηλαδή. Επισκόπηση. Οι υπηρεσίες δεδομένων και φωνής σημείωσαν τεράστια αύξηση και θέλω να αναφέρω εδώ ιδίως την αύξηση από το πρώτο έτος στο δεύτερο έτος στο Ρομιλεκτ Χομ. Home. Έχοντας ε, κατά νου ότι η πορεία που ακολουθήθηκε, η ε, καθοδική πορεία στις τιμές, δείχνει μείωση 20%, η αύξηση στη χρήση είναι 100%. Έτσι λοιπόν ο κανονισμός, και θα φτάσω σε αυτό αργότερα, είναι εντελώ αναποτελεσματικός. Γιατί είναι αναποτελεσματικός, είδαμε την παρουσίαση της Μπέρεκ, ότι έχουμε τιμές χονδρικής που είναι κάτω από τις ρυθμισμένες τιμές και για το λόγο αυτό Θέλω να σας εξηγήσω έναν όρο που λέγεται Unilateral Buyer, μονομερής αγοραστής στον κλάδο. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, έχετε μία εταιρεία στην Αυστρία και μία εταιρεία στη Γερμανία. Και αν η εταιρεία της Αυστρίας στείλει ένα πελάτη στη Γερμανία, τότε θα χρησιμοποιήσει την περιεγωγή και αντίστροφα. Και αν ε, η κίνηση ε, των δεδομένων είναι στο ίδιο επίπεδο, μιλάμε για ισορροπημένη κίνηση, για ισορροπημένη κυκλοφορία δεδομένων. Δηλαδή, το ίδιο ποσό πληρώνει ε, η εταιρεία στην Αυστρία, στην εταιρεία στη Γερμανία και συμβαίνει. Αλλά κατόπιν έχουμε ανισορροπία στην κυκλοφορία, δηλαδή όταν έχουμε μονομερή κυκλοφορία μόνο από τη μία χώρα στην άλλη και προστίθεται ε, σε αυτή την μη κυκλοφορία και δημιουργεί πολλές ε, οριακές και χαμηλές τιμές. Και αυτή η εμπορία μπορεί να γίνει μόνο αν εκπροσωπήσει και στις δύο πλευρές με δίκτυο. Αν μπορείς να προσφέρεις δίκτυο στους ε, πελάτες περιεγωγής ε, και αν θα ξεπερθούν οι πελάτες σε άλλη χώρα. Αυτή η κυκλοφορία την χάνει εμπορίου και δημιουργείται μεταξύ των ε, φορέων εκμετάλλευσης. Για να δούμε, όμως εδώ δεν υπάρχει δίκτυο, χρησιμοποιούμε ένα δίκτυο. Ε, στην Αυστρία εμείς είμαστε NBVO, φυσικά στέλνουμε πολλούς ε, πελάτες σε άλλες χώρες που χρησιμοποιούν την περιεγωγή στο δίκτυο και καθώς δεν έχουμε τίποτα με το οποίο να μπορούμε να εμπορευτούμε. Πάντοτε χρεωνόμαστε στα αριθμισμένα ανώτατα όρια. Δεν πουλάμε ικανότητα, επομένως ε, δεν μπορούμε ε, να προβούμε σε εμπόριο. Και τι σημαίνει αυτό. Το είδατε και στην έκθεση Μπέρεκα αλλά για να συνοψίσω, οι πραγματικές τιμές που πληρώνετε είναι πολύ πιο κάτω από τα ρυθμισμένα ανώτατα όρια χονδρικής και αυτό δημιουργεί τεράστιο ε, μειονέκτημα ε, για τους MVNOs. Και να έχετε κατά νου ότι σε αυτόν τον υπολογισμό που βλέπετε τις μέσες πραγματικές τιμές, Υπάρχει εδώ ε, μία ανάμειξη μεταξύ της ισορροπημένης και μη ισορροπημένης κίνησης και στην ισορροπημένη κίνηση κυκλοφορία που πληρώνεται και από τις δύο πλευρές. Αυτό δεν μετράει. Έτσι λοιπόν οι πραγματικές διαφορές μεταξύ της μη ισορροπημένης κυκλοφορίας ε, που τιμολογούνται πολύ πιο κάτω από αυτό που μπορείτε να δείτε εδώ, αλλά ακόμη και στην αξιολόγηση της Μπέρεκ κατά μέσο όρο οι τιμές που πρέπει να πληρώσουμε εμείς ως MVNO είναι 50% υψηλότερη από αυτό που πλήρωσαν μεταξύ τους οι φορείς εκμετάλλευσης. Έτσι λοιπόν τώρα σας δείχνω ένα γράφημα για το τι συνέβαινε με την περιαγωγή εντός ε, της βάσης των συνδρομητών. Εδώ βλέπετε τι συνέβη πριν και μετά την έρεξη του Rome at Home, να εξακολουθεί να υπάρχει, ε, να υπάρχουν κάποια έσοδα, γιατί έχουμε και τιμολόγηση μονάδα και σε εθνικό επίπεδο αλλά και στην περιεγωγή, αλλά μετά σας δείχνω και το κόστος που προέκυψε πριν το Rome Light at Home, είχαμε ένα μικρό περιθώριο, αλλά μετά το Rome at Home έχουμε τεράστια απώλεια. Στο τρίτο τρίμηνο βλέπετε ότι φτάσαμε σε απόλυση σε 690.000 ευρώ και αυξήθηκε αυτό σε 900.000 ευρώ στο ε, τρίτο τρίμηνο του 18. Έτσι λοιπόν ε, προσπαθήσαμε να μειώσουμε κατά 20% τις τιμές ε, χονδρικής Συνοψίζοντας, για ε, πέντε τρίμηνα πριν και μετά το Romulet at Home έχουμε 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίω σε απώλειες και αυτό αντιστοιχεί στο 20% του εργητή και στο 40% ε, του καθαρού μας κέρδους. Ποια είναι λοιπόν τα καταληκτικά μου σχόλια και το τελικό μου μήνυμα. Εμείς ως MVNOs είμαστε η δύναμη που φέρει καινοτομία μίσου των τιμών και ανταγωνισμό σε πολλές χώρες. Μας αρέσει το Rome at Home γιατί ταιριάζει απόλυτα με τις προτάσεις μας. Το καλωσορίζουμε και το καλωσορίζουν και οι συνδρομητές και ουσιαστικά συνάδει με το όραμα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Ποτέ δεν ήταν επιλογή για μας να έχουμε τιμές χωρίς ε, roaming ή για την ρήτρα ε, βιωσιμότητας και να έχουμε πρόσθετο τέλος ε, στο roaming. Δεν θεωρούμε ότι έτσι είμαστε ανταγωνιστικοί στην αγορά. Αν διατηρήσουμε αυτό το καθεστώς ως έχει υπάρχουν μεσοπρόθεσμοι κίνδυνοι. Γιατί όπως σας έδειξα, η μείωση στα τα όρια χονδρικής ε, ξεπερνάται από την ε, χρήση και εμείς ως κινητήρια δύναμη στην τοπική αγορά αποδυναμωνόμαστε από ε, αυτή την όλη διαδικασία περιαγωγής γιατί μας δημιουργεί απώλειες. Έτσι λοιπόν, αυτό που πρέπει να γίνει κατά την άποψή μας είναι δραστική μείωση των ανώτατων ε, όριων τιμών χονδρικής ε, και να δημιουργηθεί ένας νέος μηχανισμός ε, για μείωση των τιμών σύμφωνα με τα εθνικά επίπεδα τιμών στα δεδομένα. Και για να σας δώσω μία σύγκριση, εδώ βλέπετε την εφιστάμενη επιτοτική τάση. Έγινε μία αξιολόγηση το 2013 για την ε, συγχώνευση των δύο εταιριών, ε, για το πώς θα τεθούν ε, τα επίπεδα τιμών εθνικά. Και πριν πέντε χρόνια, ακόμη και τότε, το 2013, όταν μιλούσαμε για πολύ μικρότερη χρήση του 3G, η τιμή για ένα γιγαπάιτ τέθηκε στο 1,7 ευρώ. Και Μιλάμε για ένα επίπεδο το 2022 10 χρόνια αργότερα, όπου έχουμε εντωμεταξύ έκρηξη στην βιομηχανία, που είναι υψηλότερο από αυτό που είχαμε θεσπίσει το 2013. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπουμε λοιπόν ότι ήταν πολύ περιεκτικά αυτό που μας είπατε. Θα περάσουμε στον επόμενο ομιλητή, τον David Martin από την BEUC. Για να ακούσουμε την άποψή του για την κατάσταση στην αγορά αυτή τη στιγμή. Και πρωτού του δώσω το λόγο, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τη στήριξη που μας δείχνει ο οργανισμός του στο έργο μας. Έχετε το λόγο. Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, εισαγωγή σας, για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να συνεισφέρω όσο μπορώ. Από την αρχή σας είπα ότι η περιαγωγή είναι ε, ενδεικτική του τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για τους πολίτες της. Παλιά όταν ταξίδευες ε, έκλεινε, άνοιγες το κινητό σου και ευχόσου να μην σε πάρει κανείς τηλέφωνο γιατί στο τέλος του μήνα θα σου ερχόταν λυπητερή. Όμως βλέπουμε ότι τώρα ζούμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου μπορούμε να ταξιδέψουμε ελεύθερα, χωρίς ε, ε, χρεώσεις και αυτό φάνηκε από αυτά που ακούσαμε. Και φαίνεται ότι οι καταναλωτές έχουν αγκαλιάσει και υποδεχτεί θερμά τον κανονισμό Rome Like at Home. Και ήταν καιρός να γίνει κάτι τέτοιο, διότι μια ψηφιακή ενιαία αγορά πρέπει να λειτουργεί προς όφελος των πολιτών της. Και θα το ξαναπώ ότι η περιαγωγή είναι μια επιτυχία τόσο για τους καταναλωτές όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω πως μπορούμε να αισθανόμαστε υπερήφανοι για τα όσα έχουμε επιτύχει, διότι χρειάστηκε πολλής χρόνος και μεγάλη προσπάθεια από όλους, από τα θεσμικά όργανα, από τους ε, εμπλεκόμενους φορείς, από την ε, βιομηχανία και πρέπει λοιπόν να μην επαναπαυόμαστε, να βελτιωνόμαστε συνέχεια, να δούμε τι προκλήσεις ε, επιμένουν και πώς θα τι αντιμετωπίσουμε και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα, βλέπουμε ότι έχουν ε, προκύψει προκλήσεις για τα ανώτατα όρια χονδρικής και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δεδομένων αυτών λοιπόν θα ήθελα να εστιάσω σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι η πολιτική δίκαιης χρήσης και το δεύτερο σημείο τα ανώτατα όρια στις χονδρικές ε, πωλήσει. Έχουμε αναφέρει από την αρχή ότι είναι κάπως υπερβολικοί οι κανόνες. Γι' αυτό λοιπόν ε, αν η εκτελεστική πράξη χρειαστεί να αναθεωρηθεί θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι κανόνες ε, χρήζουν απλούστευσης. Και ο στόχος είναι φυσικά να μην ε, ζημιωθούν οι καταναλωτές, οι τελικοί χρήστες. Έχουμε πληροφορίες από τα κράτη-μέλη για περιπτώσεις κατάχρησης ε, της πολιτικής δικαιής χρήσης, όμως σίγουρα δεν είναι κάτι που δεν διορθώνεται. Σε ό,τι αφορά τα ανώτατα όρια στις χοντρικές πωλήσει, νομίζω πως είναι σαφές ότι αυτό είναι βασικό για να διατηρηθεί η βιωσιμότητα του όλου συστήματος και για να διατηρηθεί ο ανταγωνισμός στην αγορά. Ε, και φυσικά, ανταγωνισμός της αγοράς ε, σημαίνει μεγαλύτερες και περισσότερες επιλογές για τους καταναλωτές, καλύτερες τιμές, γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό. Το ανώτατο όριο στη χονδρική θα μπορούσε να είναι χαμηλότερο. Για παράδειγμα, διαβάζουμε στην έκθεση του Κοινοβουλίου της Επιτροπής Ήτρε που δημοσιεύτηκε πρόσφατα ότι αν συγκρίνουμε τα ενότατα όρια με το πραγματικό κόστος υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις τα ανώτατα όρια είναι σε ορισμένε περιπτώσει 10 φορέ μεγαλύτερα από τα, το πραγματικό κόστο. Είναι διαφορετικά λοιπόν αυτά που σα λέω από αυτά που ακούσατε στην προηγούμενη παρουσίαση. Αυτά τα ανώτατα όρια δημιουργούν προβλήματα ε, στου φορείς εκμετάλλευση κινητών δικτύων στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε πω πρέπει να αναθεωρηθεί η ε, νομοθεσία αυτή, η πρακτική αυτή και να κατέβουν τα ανώτατα όρια. Θα μπορούσα να συνεχίσω και να πω πάρα πολλά για το πόσο έχει υποφελήσει η περιαγωγή τους καταναλωτές. Θα περιοριστώ όμως το να πω ότι το εγχείρημα στέφθηκε με επιτυχία και πρέπει να συνεχίσουμε την επιτυχία αυτή. Άκουσα μια ερώτηση για το αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποχωρήσει από την αγορά και να την αφήσει να αυτορυθμιστεί. Νομίζω πως δεν θέλουμε να επιστρέψουμε σε καταστάσεις του παρελθόντος, γιατί όλοι θυμόμαστε τι συνέβη. Αυτό που πρέπει να κάνουμε σήμερα είναι πρώτον, αφού αισθανθούμε υπερήφανοι, να συνεχίσουμε την καλή δουλειά. Να δούμε τα προβλήματα που υπάρχουν στον ανταγωνισμό της αγοράς και να προσπαθήσουμε να μην χαθούν τα δικαιώματα που έχουν οι καταναλωτές. Ας κοιτάξουμε λοιπόν το θέμα με τα ανώτατα όρια, διότι εξελίσσεται σε μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να ευθυγραμμιστεί το κόστος δεδομένων με τα ανώτατα όρια. Θεωρώ λοιπόν ε, προσωπικά πως ε, αυτό είναι το σημαντικότερο. Θα σταματήσω λοιπόν εδώ και θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας με μεγάλη χαρά. Ε, δεν χρησιμοποίησα όλο το χρόνο που είχα στη διάθεσή μου για να μείνει περισσότερη ώρα για συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν και σας παρατηρούμε να συνεχίσουμε την καλή συνεργασία για τους καταναλωτές. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκτιμούμε πολύ το ότι κατά τη διάρκεια της Αυστριακής Προεδρίας το 2006 ξεκίνησε η δουλειά για το φάκελο αυτό και τώρα πάλι επί Αυστριακής Προεδρίας ε, ολοκληρώνουμε. Φαίνεται λοιπόν πως ε, έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος Πολλοί έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία λήψη αποφάσεων και ε, έχω πάρα πολλούς που έχουν ζητήσει το λόγο και θα δώσω τον λόγο στην ε, Πέτρα πρώτα. Δεν είμαστε και πολλοί εδώ, αλλά εμείς που ε, βρισκόμαστε εδώ, ασχολούμαστε επί με το θέμα. Ξέρω ότι ο πρόσωπο της ε, Μπέρκ μας ε, μίλησε για την περιαγωγή. Ίσως δεν υπάρχει και μεγάλη επίπτωση από πλευράς της Μπέρκ. Η Μπέουκ ζήτησε τα εθνικά μέλη να προβούν σε μία διαφανή τιμολόγηση και νομίζω ότι υπάρχει ευαισθητοποίηση του καταναλωτή ως προς τη χρήση. Συμφωνώ με τις επιχειρήσεις ότι έχουν δυσκολία να πουλήσουν κάτι αν οι καταναλωτές ε, δεν προτίθενται να το χρησιμοποιήσουν ως υπηρεσία. Αυτή είναι η ευρεία εικόνα. Σας ευχαριστώ πολύ για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις. Αυτό το παλαιό έγγραφο ε, που το βλέπετε ε, μιλούσαμε για 8,5 γίγκα και βλέπετε τα, το αποτέλεσμα στο MVNO. Αλλά η Επιτροπή είχε προτείνει 8,5 ευρώ ανά γιγκαμπάιτ. Αυτή ήταν η αρχική πρόταση. Αν είχατε ακούσει το Κοινοβούλιο, τότε θα μιλούσαμε για 3 ευρώ ανά γιγκαμπάιτ και 1 ευρώ το 2022. Αυτό ήταν, αυτή ήταν η έκβαση του τριμερούς διαλόγου, όπου το Συμβούλιο είχε αρχίσει από 10 ευρώ και η έκβαση είναι ήταν αρχίζοντας από 7,7 ήμασταν στα 6 και σε 1,5 μήνα στα 4,5 ευρώ. Αν νομίζετε ότι σφάλουμε, και ότι θα έπρεπε να είχαμε ακολουθήσει τους επιχειρηματίες, τους παρόχους, την Κομισιόν ή το Συμβούλιο, καταλαβαίνετε ότι θα ήταν ε, εντελώς διαφορετικό το αποτέλεσμα. Εγώ εργάστηκα ε, από την πλευρά μάλλον του ανταγωνισμού. Φυσικά οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται και για τον ανταγωνισμό, αλλά και για τις επενδύσεις που χρειαζόμαστε. Τώρα, το μεγάλο ερώτημα είναι το εξής. Όπως είπε και η ομιλήτρια, η κυρία Φούρ, χρειάζονται επενδύσεις και υπάρχουν. Μιλάμε και για τις επενδύσεις για το όλο φάσμα. Βλέπουμε την πρώτη έκβαση του 5G. Στην Ιταλία πληρώνει κανείς πέντε φορές περισσότερο από ό,τι στη Φιλανδία. Πώς λοιπόν θα φτάσουμε σε μία ψηφιακή ευρωπαϊκή αγαρά τη στιγμή που δεν καταβάλλονται τα χρήματα ε, αναχώρα όπως θα έπρεπε. Αυτό δεν το δέχτηκαν ε, τα κράτη-μέλη, δεν ε, δέχτηκαν την αντιστάθμιση τα κράτη-μέλη, αλλά ξέρετε ότι το επόμενο βήμα στο επόμενο βήμα, αν πληρώσει κανείς για το φάσμα, για όλο το φάσμα, ποια θα είναι η χρήση του. Γιατί υπάρχει αυτή η τεράστια διαφορά. Στην Αυστρία 220 MB ετησίως είναι η χρήση του φάσματος. Στη Φιλανδία είναι το διπλάσιο. Αν σας ενδιαφέρει η Γερμανία, είναι το 1 δέκατον του φάσματος χρήσης από την Αυστρία. Τη στιγμή που πληρώνουν οι επιχειρήσεις για το φάσμα, μετά δεν χρησιμοποιείται. Και τότε δεν θέλουν άλλοι να έχουν ευθυνή πρόσβαση στο φάσμα. Άρα υπάρχει περισσότερη αγορά, δηλαδή μπορούμε να εμβαθύνουμε αλλά αυτή η αξιολόγηση χρήσης του φάσματος δεν μας οδήγησε πουθενά. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει follow-up από την Κομισιόν, ζητάμε όμως μία αναθεώρηση. Αυτό το ε, αναφέρω, φωνάζω γι' αυτό εδώ και χρόνια, γιατί δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη χρήση του φάσματος τη στιγμή που βλέπουμε ότι δεν αλλάζουν οι τιμές. Γιατί δηλαδή χρησιμοποιείτε το φάσμα κατά διαφορετικό τρόπο αναχώρα. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ωραία. Άλλοι που θα ήθελαν το λόγο. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει εξισορρόπηση, γιατί δεν μιλάμε για μια, μικρό και, για μια μικρή χώρα και ένα μικρό πάροχο, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει ανισομέρεια και ανάμεσα μεγάλων χωρών, δηλαδή αυτοί που δεν έχουν την ιδιοκτησία του δικτύου, στέλνουν προς τα έξω αυτές τις παροχές, αλλά δεν τις παίρνουν πίσω. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η ανισομέρεια. Και τα μέλη της Μπέρεκ το ανέφεραν αυτό, ότι δεν είναι εύκολο αλλά όταν το έχουμε, τότε μπορεί να γίνει ευρεία χρήση του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση. Ελπίζα ότι θα ήταν εύκολη, αλλά τελικά μπορεί να αποδειχτεί και πολύπλοκη. Γιατί ήταν απαραίτητο να έχουμε ένα τέτοιο διοικητικό μέτρο τόσο χωροκατακτητικό, γιατί οι αγορές ε, δεν έλαβαν μόνες τους τα μέτρα αυτά. Οι εταιρείε ήξεραν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι οι πελάτες ε, με τις χρεώσεις της περιεγωγής Όποτε ταξίδευε κανεί ε, στο εξωτερικό, σήμαινε ότι έπρεπε να ξοδέψει πολλά χρήματα στο τηλέφωνο. Γιατί αυτό λοιπόν έπρεπε να λυθεί με νομοθετικά μέσα. Γιατί οι δικές σας ε, εταιρείε δεν έκαναν το ίδιο από μόνες τους. Γιατί χρειαζόταν ε, να τους αναγκάσει το κοινοβούλιο να το κάνουν αυτόν, αν μπορώ να το θέσω με αυτά τα λόγια. Γιατί λέτε τώρα ότι έχει αυξηθεί ο κύκλος εργασιών, έχει αυξηθεί η χρήση. Έτσι λοιπόν, από οικονομική σκοπιά, αυτό που συνέβη ήταν πολύ καλό. Λαμβάνοντας αυτού, εμείς που ήμασταν ε, σκιώδεις εισηγητές, αλλά και ο ίδιος ο εισηγητής ε, πέρασαν ε, από πάρα πολύ δύσκολες συζητήσεις με τις εταιρείες οι οποίες παρουσίαζαν σενάρια καταστροφής. Γιατί λοιπόν οι εταιρείε δεν το έπρεξαν αυτό από μόνο του και να δράξουν όλα τα ωφέλη τα οποία υπάρχουν τώρα. Νομίζω ότι και την επόμενη φορά πάλι θα πρέπει να παρέμβουμε. Και πάλι θα πρέπει να ρυθμιστεί αυτό με διοικητικά μέτρα. Και ξέρουμε ότι αυτό θα αποτελέσει τεράστια ευκαιρία για την αγορά. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι γιατί θα πρέπει κάθε φορά να παρεμβαίνει η νομοθετική αρχή. Εγώ έχω μιλήσει με πολλές εταιρείες και ε, εγώ έχω ε, ουσιαστικά ιστορικό σε τεχνολογίες πληροφοριών ε, και γιατί, παραδείγματος χάρη, στην Γερμανία ή στην Τσεχία οι εταιρείε λένε αν καταργείται το roaming θα υπάρχει τεράστιο κόστος για μας. Εγώ ε, νομίζω ότι δεν υπήρξε κόστος ε, γιατί ήταν όλα σε ένα σερβερ και έτσι λοιπόν σε ό,τι με αφορά θέλω να είναι οι εταιρείε τηλεπικοινωνιών φιλικές προς το χρήστη έτσι ώστε να μην χρειάζεται να περνάμε από αυτή την ε, δυσάρεστη νομοθετική διαδικασία. Ναι, υπάρχει τεχνικό κόστος, αλλά πάνω κάτω το κόστος αυτό είναι το ίδιο σε όλη την Ευρώπη. Δεν νομίζω υπάρχουν τεράστιες διαφορές ε, μεταξύ Τσεχίας, Ιταλίας, Φιλανδίας. Υπάρχει λοιπόν επιθυμία από τη δικαιωτικού σας οργανισμούς να είστε πιο φιλικοί προς το χρήστη. Ίσως να είναι δύσκολη η ερώτηση που σας έθεσα. Σας παρακαλώ. Ε, σας ευχαριστώ πολύ, κύριος Κόλιτσεκ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσα να μιλήσω ισπανικά, αλλά τελικά θα μιλήσω τσέχικα, γιατί είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, ρώτησε ο συνάδελφος γιατί πρέπει να αναγκάσουμε τις εταιρείες τηλεπικοινωνίων να κάνουν κάτι που τελικά είναι προς όφελός τους, ό,τι αφορά τις μεγάλες εταιρείες. Ποιος είναι ο αντίκτυπος αυτού που ξεκινήσαμε εδώ. Δηλαδή, συγκεκριμένα να έχουμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δίκτυο ίντερνετ υψηλών ταχυτήτων. Και αναρωτιέμαι αν ο κύριος Κράμερ θα μπορούσε να μου πει σε ποιο βαθμό αυτή είναι μια σημαντική ευκαιρία και για αυτούς ε, ως ε, φορείς εκμετάλλευσης ιδεατών δικτύων. Ευχαριστώ. Ωραία. Θέλει άλλο το λόγο. Δεν βλέπω κάποιον άλλο. Ποιος ε, θέλει να ξεκινήσει. Να ξεκινήσουμε τον κύριο Κράμερ και να το κάνουμε αντίστροφα. Παρακαλώ. Αν κατάλαβα καλά, θέσατε την ερώτηση γιατί χρειάζεται η ρύθμιση της αγοράς για την περιεγωγή. Νομίζω ότι ο κύριος Ρούμπιχ μπορεί να απαντήσει στην εντέλεια, γιατί παρακολουθεί το ιστορικό για τις τιμές περιεγωγής εδώ και καιρό. Από τη θέση ενό φορέα εκμετάλλευση και λειτουργώντας ως φορέας εκμετάλλευση στις αγορές εδώ και 20 χρόνια, πάντοτε είμαστε με δύναμη στην αγορά, ως υπεύθυνος διευθυντής μιας τέτοιας εταιρείας, πάντοτε σκέφτεσαι που θα μπορούσε να είναι το ανταγωνιστικό σου πλεονέκτημα. Είναι καλύτερο να έχεις χαμηλές ιατρικές τιμές με κόστος ε, σε υψηλότερες τιμές ε, στην περιαγωγή το αντίστροφο και απεδείχθη τουλάχιστον στην Αυστρία και στη Γερμανία ότι οι χαμηλότερες εθνικές ε, τιμές είναι ε, ουσιαστικά ένα καλύτερο επιχείρημα για να έχουμε νέους συνδρομητές και να διατηρήσουμε τον αριθμό των συνδρομητών. Βέβαια, υπήρχε μια ειδική αγορά, ε, υπήρχε ανάγκη για ε, υπηρεσίες περιαγωγής σε συγκεκριμένα τμήματα και προσφέραμε ειδικές τιμές για την περιαγωγή. Αλλά, εδώ και χρόνια, Πάντοτε ήμουν οπαδός μιας ρύθμισης ε, για την ε, χονδρική για να δώσουμε και στους ε, MNOs αλλά και στους VMNOs να μπουν σε αυτό το τμήμα. Έτσι, λοιπόν, κατάλαβα ότι η απόφαση ήταν αντίστροφη, την καταλαβαίνω και τη δέχομαι. Η απόφαση ήταν να έχουμε ρύθμιση και στο επίπεδο λιανικής και χονδρικής έγινε και το έχουμε τώρα και ο κανονισμός είναι rom Late at Home ε, θα μπορούσε να είναι πιο εύκολο για τους καταναλωτές αν το καθεστώς ε, χονδρικής ε, είναι σωστά και αυτό μπορεί να είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και αυτή ήταν η ερώτησή σας θα μπορούσε να είναι πολύ καλή ευκαιρία για τους μικρούς φορείς εκμετάλλευσης αν είχε γίνει σωστά. Δηλαδή, αν βάλετε τις τιμές χονδρικής επίπεδο κόστος, ε, τότε θα δείτε ότι οι μικρότεροι φορείς εκμετάλλευσης και οι MVNOs ε, θα αφαιρέσουν πιθανότατα τη ρήτρα της δικής χρήσης, γιατί πάντοτε ε, ουσιαστικά βλέπουμε μείωση της της πολιτικής. Ε, Τη δικής χρήση. Τώρα έχουν βελτιωθεί πολύ τα πράγματα σε σύγκριση με το παρελθόν για του καταναλωτέ, αλλά δεν είναι τέλεια κατάσταση. Εξακολουθεί να υπάρχει σύγχυση. Έχεις ε, κάποιες τιμέ χωρίς περιαγωγή και αν ε, βάλεις όλες τις προσπαθίες σου στις τιμέ, τελικά πά σε μια άλλη χώρα και δεν μπορεί να έχει περιαγωγή πια. Άλλο είδη τιμών που σου προσφέρεται είναι ότι ε, συνεργάζεσαι με φορείς που έχουν την τρεφησιμότητα, έχει το fair ε, τη δίκαιη χρήση και μετά έχει κάποιες τιμές που αντιστοιχούν στο ROM Light at Home ε, με απεριόριστη κατανάλωση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποια μεγάλα βήματα έχουν γίνει λοιπόν, αλλά το τελικό βήμα πρέπει ακόμη να γίνει. Thank so Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Φουρ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σε ό,τι αφορά το... τους χρήστες και το εύρος ε, και το φάσμα, ε, είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε μια σύγκριση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα στη Φιλανδία είναι διαφορετικά τα πράγματα, διότι εκεί χρησιμοποιείται η κινητή τηλεφωνία κατά πολύ. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή στο πώς αξιολογούμε τα δεδομένα αυτά. Νομίζω ότι με το 5G το κόστος του φάσματος ε, θα αλλάξει διότι θα χρησιμοποιούμε ε, περισσότερο, περισσότερες συχνότητες. Ε, τώρα, δεν χρειάζεται να πάρουμε τόσο παραμυθατικά μέτρα. Θα έλεγα μάλιστα πως δεν χρειάζεται. Η αγορά εξελίσσεται, υπάρχει υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού Και είδαμε μία περίπτωση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ρύθμισε μία αγορά στην οποία ο ανταγωνισμός είναι αρκετά υψηλός και από ό,τι μας πληροφόρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε αυτή την περίπτωση στην κινητή τηλεφωνία υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Το Roam Like at Home μπορεί να αύξησε τον όγκο ε, χρήσης, δεν αύξησε όμως τα έσοδα. Και αν κοιτάξουμε τα ανώτατα όρια τιμών, τα οποία έχουμε ήδη συζητήσει πολύ, και το θέμα των φορών εκμετάλλευσης ε, δικτύων, θα δούμε ότι η αγορά κινητών δικτύων είναι αρκετά ενεργή. Έχει γίνει λοιπόν και η ανάλυση που έχει γίνει, έχει γίνει σε δύο χώρες και όχι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο κύριος Κράμερ είναι Αυστριακός, οπότε μας ε, παρουσίασε τη δική του εμπειρία από την Αυστρία. Όμως υπάρχουν διαφορές και από κράτος κράτος και από αγορά σε αγορά και από τον κλάδο στον οποίο κινείται κανείς. Εγώ εργάστηκα 10 χρόνια ε, στον χώρο των πωλήσεων ε, φορών εκμετάλλευσης κινητών δικτύων στην Δανία. Και εκεί είχαμε άλλες ε, προκλήσεις. Υπήρχαν φορείς που ήθελαν να μπουν στην αγορά και δεν μπορούσαν λόγω των ετοιμών. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν φορείς εκμετάλλευσης οι οποίοι κινούνται στην ε, αγορά και είναι αρκετά ισχυρή. Η αγορά μας είναι λοιπόν πολύ ανταγωνιστική. Ε, τώρα, δεν θα γυρίσουμε πίσω, διότι τα δίκτυα υπάρχουν. Υπάρχουν ε, φορείς όπως η Vodafone, για παράδειγμα, που έχουν τα δικά τους δίκτυα. Η δημιουργία ανώτατων των ορίων και σε συνδυασμό με τιμές που βρίσκονται πολύ χαμηλότερα από αυτή είναι, θεωρώ, κάτι το φυσιολογικό. Δεν βρίσκω ούτε στην έκθεση της Μπέρεκ, ούτε στην έκθεση της Επιτροπής Ήτρε κάποιο ε, ακλόνητο επιχείρημα υπέρ της ε, περαιτέρω ρύθμισης της αγοράς. Ας θεωρήσουμε το Rome Like at Home επιτυχία και ας εστιάσουμε στα πλεονεκτήματα που αυτός ο κανονισμός ε, επέφερε στους χρήστες. Σίγουρα έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας, όμως έχουμε και μια νέα πραγματικότητα που έρχεται. Υπάρχει το 5G, σύντομα θα είναι παντού. Αν πιέσουμε ακόμα περισσότερο την αγορά θα βάλουμε σε κίνδυνο τις επενδύσεις στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι οι επενδύσει ε, στι ΗΠΑ είναι διπλάσια σε σχέση με τι επενδύσει στην Ευρώπη. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή διότι η αγορά είναι δύσκολη, είναι περίπλοκη και οποιαδήποτε ρυθμιστική παρέμβαση από εμά θα επηρεάσει όλους και όχι μόνο τις ε, επιχειρήσεις αλλά και ε, την ταχύτητα ε, με την οποία θα αναπτυχθεί το 5G αλλά και τα δίκτυα τα ίδια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κότφερ έχει το λόγο. Νομίζω πως δεν έχω να σχολιάσω πολλά, μόνο δύο σχόλια. Γιατί λοιπόν χρειάζεται... Γιατί εφόσον δεν χρειαζόταν να αναλυφθεί δράση από το Κοινοβούλιο και από την νομοθεσία, γιατί έγινε. Βλέπουμε το φάσμα πως, ε, της αγοράς ε, ότι είναι πάρα πολύ ε, διαφορετικό. Βλέπουμε ότι μεγάλη φορούς εκμετάλλευση είναι λίγοι, είναι το πολύ τέσσερις. Επηρεάζουν λοιπόν με αυτό το ολιγοπόλιο την αγορά. Πριν ακούσω να πω ότι πριν τις ε, παρεμβάσεις οποιοδήποτε πάροχος υπηρεσιών υπολόγιζε το κόστος παροχής υπηρεσιών στην εγχώρια αγορά και στην ε, αγορά του εξωτερικού διαπίστωνε ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές στις τιμές και φυσικό επόμενο ήταν αυτές, αυτή η διαφορά να αντικατοπτρίζεται και στις ε, τιμές. Όμως, ό,τι αφορά τι χονδρικέ πωλήσει, ο ανταγωνισμό ε, της αγοράς έχει οδηγήσει στην μείωση ε, των τιμών. Περαιτέρω μείωση θα είχε πολλά προβλήματα. Κυρίως ε, για το ότι δεν θα κατάφερναν να αυξήσουν το πελατολόγιο και τον, και τον όγκο των δεδομένων, γιατί όταν ε, κάνει συμβόλαιο με μια εταιρεία παροχής κινητής τηλεφωνίας, ε, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι σίγουρα δεν είναι η περιαγωγή. Ο ανταγωνισμός και μόνο δεν θα οδηγήσει στην ε, πτώση των ε, τιμών. Γι' αυτό και έχει αποδειχθεί ότι έπρεπε να υπάρχει κάποια παρέμβαση νομοθετική. Βέβαια, τώρα το τι θα μπορούσε να είχε γίνει ε, είναι μια άλλη ερώτηση. Αλλά η Μπέρεκ τα επόμενα χρόνια θα έχει πολύ δουλειά να κάνει έτσι ώστε η εφαρμογή του νέου κανονισμού να γίνει ομοιόμορφα. Επίσης έχουμε εστιάσει σε ανάπτυξη νέων στρατηγικών και σε κάποιες έρευνες που θα δώσουν απάντηση στα ερωτήματα που θέσατε αρκετοί από εσάς εδώ. Και καταρτίζουμε προγράμματα για το 2020 και μετά. Και εδώ η συνεισφορά σας είναι πολύτιμη. ευχαριστούμε πολύ. Και τέλος ο τελευταίος μας ομιλητής. Ευχαριστώ. Νομίζω ε, όταν δείτε την αγορά τηλεπικοινωνιών, λέει ο David Μάρτιν από τη Μπιούκ, οι αγορές βαίνουν καλώς για τους καταναλωτές, γιατί είναι σε μια ευάλωτη θέση και γι' αυτό θα πρέπει να ρυθμίσουμε τις αγορές με τον κανονισμό περι, περιαγωγής έτσι ώστε οι καταναλωτές να έχουν μια καλή υπηρεσία σε δίκαιη τιμή. Ε, δεν κατανοούμε πάντα αυτές τις προσφορές από τους παρόχους. Δυστυχώς τώρα γιατί δεν αυτορυθμίστηκε η αγορά. Έχω την εντύπωση ότι ολόκληρη η αγορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο λειτουργούσε σαν καρτέλ, διότι όλοι ευεργετούνταν από το συμπληρωματικό τέλος περιαγωγής, άρα ήταν σαφές ότι δεν θα ήθελαν να χάσουν αυτό το κέρδος από μόνες, τις, από μόνες τους οι επιχειρήσεις. Θα πρέπει να είμαστε πιο φιλικοί προς τον καταναλωτή. Βεβαίως, εάν κανείς πληγεί ως προς την ε, πηγή βασικού κέρδους. Σκεφτήκαμε και σκεφτόμαστε ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει το προβάδισμα, να παρέμβει δηλαδή γιατί αυτό ακριβώς σημαίνει ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, ψηφιακή αγορά, κάτι το οποίο είναι ουσιώδες ως προς την οικοδόμηση της Ένωσης. Άρα, αυτοί οι κανόνες είναι τόσο σημαντικοί όσο ήταν και στο παρελθόν και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα για να φτάσουμε στον απότερο στόχο, δηλαδή την απαλυφή όλων αυτών των ε, συμπληρωματικών τελών και να προωθήσουμε τον ανταγωνισμό υπέρ των ε, καταναλωτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ζητήσουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει τι ε, αποκόμισε από την ακρόαση, ποιο θα ήταν το μέλλον της περιαγωγής και τι θα γίνει στις 13 Ιουνίου 2022 που λύγει ο κανονισμός και τι θα γίνει για την παγκόσμια ε, περιαγωγή. Τι θα γίνει ε, σε σχέση με τις διμερείς συμφωνίες με την ITU, ε, με τον Οργανισμό Διεθνών Τηλεπίδρασης Επικοινωνιών. Τι θα κάνει η κυρία Μάλμστρομ, διότι μας είπαν ότι το roaming πρέπει να βασίζεται σε ένα τίμημα. Θα θέλαμε να δούμε τι κάνει η κυρία Βεστάγκερ. Παρακολουθεί τις εξελίξεις. Συζήτησα ε, με τον κύριο Βιόλα, τον Γενικό Διευθυντή και μου είπε ότι το 2007 ήταν η πρώτη φορά που μας ε, απασχόλησε η περιαγωγή και το κόστος της. Άρα έχουμε εξελίξεις αναπάνταχες. Εγώ μία εβδομάδα πριν ήμουνα στην Κίνα όπου συζητήσαμε για την τεχνητή νοημοσύνη και για την συλλογή δεδομένων Γι' αυτό οι τηλεπικοινωνίες θα διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να προωθήσουν και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Από την Επιτροπή έχουμε τον Αντώνη Βίλαν, Γενική, Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Connect. Τι έχεις να μας πεις, Άντωνη. Ευχαριστώ. Μπορώ να σας επιβεβαιώσω Καταρχήν ότι χαιρόμαστε που μπορούμε να παρέμβουμε και που είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε σαφή στοιχεία, αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση με την εξελισσόμενη πορεία. Όπως ξέρετε ο κανονισμός περι, περιαγωγής προβλέπει όχι μόνο συνεκτική αναθεώρηση στο τέλος του επομένου έτους, αλλά και μία ενδιάμεση έκθεση στο τέλος του έτους, το Δεκέμβριο δηλαδή. Βρισκόμαστε στα τελικά, στο τελικό στάδιο μπορούμε να αντλήσουμε πολλά σημαντικά δίδαγματα και φυσικά δεν θα ήθελα να σας αποκαλύψω το περιεχόμενο, αλλά υπάρχει συνέπεια με τα μηνύματα που ακούσαμε σήμερα, γιατί λαμβάνουμε υπόψη τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει συλλέξει η Μπέρκ μέσα στα πλαίσια της ε, πολύ σημαντικής μας συνεργασίας σε αυτό το τομέα. Ε, δεν είναι λοιπόν μυστικό το ότι θεωρούμε την ευρεία ε, χρήση της περιαγωγής και του Roam Like at Home σαν ένα μέσο για να μπορέσουν οι καταναλωτές να αντιμετωπίσουν την διωγγούμενη ζήτηση φυσικά ε, έχουμε να κάνουμε και με αριθμητικά στοιχεία που είναι εξατομικευμένα. Είχαμε και ένα μήνυμα από έναν πάροχο όπου είχαμε έκρηξη ως προς την χρήση των δεδομένων. Αλλά σε γενικές γραμμές θα ήταν ε, πολύ δύσκολο να αρνηθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Αυτό θα ήταν το ολίγιστο. Ως προς το ερώτημα του κυρίου Τοσανόφσκι, αυτό το ερώτημα είναι πολύ σημαντικό. Από την απαρχή των ε, κανονισμών περιαγωγής υπάρχει ε, μία παρέμβαση στην αγορά, η οποία όμως θεωρείται εξαίρεση. Η αγορά θα πρέπει να αυτοδιορθωθεί ή να μας δώσει στοιχεία ότι θα μπορέσει να αυτοδιορθωθεί ελήψη κανονισμού και ο Τζέρεμι Γκότφρι αυτό ακριβώς τόνισε. Όταν δούμε τις ανώτατες ε, τιμές χονδρικής, βλέπουμε ότι θα πρέπει να γίνει μια αποτίμηση της συμπεριφοράς της αγοράς και κατά πόσο συμπεριφέρεται καλύτερα σε σχέση με προγενέστερα εγχειρήματα. Ένα άλλο θέμα που αφορά τη χονδρική, τις τιμές ε, χονδρικής που ανέφεραν οι περισσότεροι ομιλητές, είναι να έχουμε ε, αξιόπιστα μέτρα ως προς τη διαχείριση του κόστους και εδώ ε, έχουμε επαφές με την ΠΕΡΚ και τους παρόχους έτσι ώστε να έχουμε ένα αξιόπιστο πρότυπο κόστους ε, της αγοράς που να συσχετίζεται με το κόστος των δικτύων. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο για την συνεκτική αναθεώρηση που θα υποβληθεί στο τέλος του επόμενου έτους. Δεν θα πρέπει να προτρέχουμε ούτε να επισπεύσουμε τα πράγματα, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν θα πρέπει ε, με περιορισμένα στοιχεία να φτάσουμε σε αναπόδραστα ε, αποτελέσματα και συμπεράσματα περισσότερο σε σχέση με τη χρήση δεδομένων. από το εύρυ κοινό. Ένα από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν και στην ενδιάμεση έκθεση και την ε, συνεκτική αναθεώρηση του επόμενου έτους είναι να δούμε πώς δρούν οι διάφοροι φορείς ε, ε, αγοράς. Όχι μόνο οι MVNO σε σχέση με τους MNO, αλλά και οι φορείς της αγοράς που λαμβάνουν περισσότερα ε, στοιχεία ή στέλνουν προς τα έξω αυτή την κίνηση δεδομένων. Αυτό θα έχει μεγάλη σημασία για να υπάρχει η εγγυήση ότι έχουμε ένα εξισορροπημένο καθεστώς ή τουλάχιστον να αναγνωρίσουμε ε, μέτρα διόρθωσης της αγοράς. Γι' αυτό και καταγράψαμε πολλά από τα επιχειρήματα που προβάλλατε σήμερα. Τέλος, το πρώτο τελευταίο μάλλον ε, σχόλιο αφορά την πολιτική δικαιοχρησίας που ανέφεραν ορισμένοι παρεμβαίνοντες. Εδώ θα πρέπει να φτάσουμε σε μία εξισορρόπηση γιατί οι κανόνες όπως ε, έχουν είναι πιο περίπλοκοι από όσο θα ήθελαν μερικοί για να προστατεύσουμε τον ε, ε, καταναλωτή και να καλύψουμε το ευρύ φάσμα συμπεριφοράς ή συμπεριφορών του καταναλωτή. Θα πρέπει να γίνουν αυτά τα αντισταθμίσματα πολλές φορές και γι' αυτό θα πρέπει να επανεξετάσουμε και το ρυθμιστικό πλαίσιο για να αποτιμήσουμε αυτούς τους κινδύνους. Τέλος, για να απαντήσω στο ερώτημα της κυρίας Γκρίφιν, ως προς το λυπηρό θέμα του Brexit, εάν δεν υπάρξει συμφωνία, η Επιτροπή οποία έχει προβάλει ε, δελτία ε, ετοιμότητας, ένα από τα οποία αφορά και τις τηλεπικοινωνίες. Στην περίπτωση, δηλαδή, στην περίπτωση όμως που υπάρξει συμφωνία απόσυρσης που υπάρχει επιτάπητος θα έχουμε μία ε, μεταβατική περίοδο έτσι ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Και τέλος, ένα προσωπικό σχόλιο. Κύριε Χούμπε, εγώ δεν είμαι στο παιχνίδι της ε, περιαγωγής ε, τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα όπως εσείς. Το 2010 όμως ε, συντάξαμε τον κανονισμό για την ψηφιακή αγορά και θεωρήσαμε ότι οι τιμές περιαγωγής μέχρι το 2015 θα συσχετιστούν με τις εγχώριες τιμές. Χρειάστηκε όμως περισσότερος χρόνος, αλλά πολλές φορές οι προβλέψεις ε, λειτουργούν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να βλέπουμε ότι το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ουσιαστικά κατευθύνει το θεματολόγιο, βάζουμε τα δυνατά μας και έχουμε και μια ιστορία επιτυχίας. Ε, σας, αν δείτε γιατί είναι σημαντική η Ευρώπη για τους καταναλωτές, ε, το roaming είναι πάντοτε κάτι που αναφέρεται είναι μια τέτοια περίπτωση. Συνεχίζουμε λοιπόν τον αγώνα, προσπαθήσουμε να βρούμε καλύτερες λύσεις. Εγώ έχω συνομιλήσει και με την Επίτροπο, τη Μαρία Γκάμπριελ, έχει δεσμευτεί απόλυτα για το θέμα αυτό και σίγουρα και η ακρόση ε, της Επιτροπής ε, θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα του χρόνου. Ε, θα δούμε τι θα κάνει και ο νέος Επίτροπος. Ε, η κυρία Κρούς ένα δεύτερο γύρο, μάλλον χρησιμοποιήσει και δεύτερο γύρο για να απαντήσει αυτές τις ερωτήσεις. Είναι ζωτικό λοιπόν να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος επίτροπος και τι μπορεί να κάνει για τους πολίτες μας και επίσης και στις ε, προεκλογικές εκστρατείε. Νομίζω ότι αυτός είναι ο θετικός τρόπος να προωθούμε τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Ολοκληρώνουμε εδώ τη συνεδρίαση. Η επόμενη συνεδρίαση μας θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου από τις 3 το απόγευμα στις 6.30 και στις 22 ε, Νοεμβρίου, σήμερα δηλαδή, ακυρώνεται η απογευματινή συνεδρίαση. Είμαστε ένα μήνα πριν τα Χριστούγεννα, σας εύχομαι τα καλύτερα. Καλά δώρα και τα λέμε στην επόμενη συνεδρίαση.